Ευχαριστώ τον εισηγητή. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι, στις 12 η ώρα. Τώρα στη συνέχεια έχουμε την έκθεση Κορνέλης Φίσερ για τη διατήρηση των λεπτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων. Η κυρία Φράγκα Εστέβε θα αντικαταστήσει τον την εισηγητή και θα το προτείνει για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο συγκριτή έχει αναφέρει κάποιε βασικέ ανησυχίε που δημιουργούνται από την πρόταση τη Κομισιόν, παραδείγματο χάρη τάση ρυθμιση αναπεριοχών θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο του κοινοτικού πυλώνα. επίση τεχνικά μέτρα. Ε, προσέγγιση που μπορεί να είναι κατανοητή, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε οι περιφερειακοί κανονισμοί να περιορίζονται σε εφαρμοστικέ μόνο πτυχέ και στη ρύθμιση τεχνικών λεπτομεριών. Και το λέω αυτό γιατί η εκπώνηση ε, των κανονισμών πλαισίου περιλαμβάνουν ελάχιστα στους ε, κανόνες και μετά πόνηση νομοθετημάτων ανατομέα με όλο και με συχνότερη προσφυγή στην επιτροπολογία είναι ένας από τους ε, τρόπους που φαίνεται να, να θέλει να εξαντλήσει η Κομισιόν εν ώψη προοπτικής ε, συναπόφαση θέματα αλίας όπως λέγεται, ε, χωρίς επιτροπές στην υπεκφυγή, στην πράσινη βίβλο τη σχετική. Δεν μιλάμε όμως για μια οποιαδήποτε πολιτική, αλλά για μια κοινή πολιτική. Άρα πρέπει να είναι σαφές τι μπορεί να συνεπάγεται μια λιγότερο ή περισσότερο εμφανής ε, εκχώρηση εξουσιών στα κράτη-μέλη. Και πρέπει να προσέξουμε ότι οι κανόνες αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν είναι να επιβάλλουν τους κανόνες και να μην δημιουργούν διακριτική μεταχείριση. Έχουμε λοιπόν τον καθορισμό κάποιων ε, μεγεθών στους περιφερικούς κανονισμούς. Αυτά τα μεγέθη αλλά και τα μέτρα, η μέτρηση των ματιών και ε, όλοι οι άλλοι σχετικοί κανονισμοί θα πρέπει να είναι κοινοί και να εγκρίνονται από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Επίσης, από αυτή την έννοια, Έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις από την Επιτροπή Αλίας σε προτινόμενες για την εφαρμογή της διαδικασίας της επιτροπολογίας σε πολύ λεπτομεριακές πτυχές. Επαναλαμβάνω, το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίζει για τις ε, περιόδους ε, ανάπαυσης, για τα μάτια των δικτυών, για τις απορρίψεις κτλ. Διότι όλοι οι κοινοτικοί φορείς θα πρέπει να τηρούν κάποιους ελάχιστους κανόνες παιχνιδιού, οι οποίοι θα είναι κοινοί για όλους. Από αυτή την κοινή πολιτική κοινοτικοποιημένη είναι μόνο η πρόσβαση στις αγορές. Ενώ η πρόσβαση ε, στην αγορά η διαχείριση αφήνουν κάποια περιθώρια ελιγμών που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη για να αποφεληθούν οι δικές, οι δικές τους σε βάρος των στόλων των άλλων κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κοινοτικοποιήσει και να αναρμονίσει τον έλεγχο. Δεν καταλαβαίνουμε όμως πώς με άλλα μέτρα τελικά γίνεται κατακαιρματισμός, διαχωρισμός και δημιουργούνται διαφορετικοί κανόνες για τον ίδιο το παιχνίδι ανάλογα με τον τόπο στον οποίο παίζεται εντό αγωγικών. Πρέπει λοιπόν να είναι αξιόπιστη η κοινή πολιτική και για να έχει το μέλλον που θα πρέπει δεν θα πρέπει να έχουμε τίποτα πριν από του 2012. Τώρα σε ό,τι αφορά το ενιαίο δίκτυο υπάρχει μία εναλλακτική οδός για το ένα ενιαίο δίκτυο, λοιπόν, αν θα πρέπει σε κάποιο σκάφος να υπάρχει περισσότερα του ενός ε, είδη ε, δικτύων. Αυτά, ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ, Επίτροπος, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ τον κύριο Φίσερ και την κυρία Φράγκα και την Επιτροπή Ελία για το σχέδιο έκθεση τη πρόταση τη Επιτροπή για τεχνικά μέτρα ε, για τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα τεχνικό ζήτημα και όπω ε, γνωρίζετε, τα τεχνικά μέτρα διατήρηση των αποθεμάτων στι περιοχέ αυτέ είναι, είναι πολύ σημαντικά και, και περιέχονται σε διάφορου κανονισμού ο γενικό ε, κανονισμό ε, τεχνικό του 1998, ο επιπρόσθετος κανονισμό για την ανάκτηση ε, των αποθεμάτων και ο τήσιος κανονισμός, ο οποίο επίση περιέχει ορισμένα μέτρα, τεχνικά μέτρα διατήρηση. Πέραν τη νομική πολυπλοκότητα, οι φυστάμενοι κανόνε σε ορισμένε περιπτώσει είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και είναι δύσκολο να, να... να ελέγχονται. Η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση για ένα νέο κανονισμό για το θέμα αυτό στο Ατλαντικό Ωκεανό 4 Ιουνίου του περασμένου Η πρόταση διατυπώθηκε μετά από εκτενείς διαβουλεύσει με του ενδιαφερόμενου και με τα κράτη-μέλη ε, κατά τη διάρκεια του 2006-2007 ε, και ομοδοποιεί όλους τους ε, σχετικούς κανόνες σε μία και μόνο νομοθετική πράξη, η οποία θα βελτιώσει την νομική συνέπεια με τον τρόπο αυτό. Επίσης, η πρόταση έχει ως στόχο την απλοποίηση και τη διασαφήνιση των διαφόρων κανόνων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην απλοποίηση ποιήση των ελέγχων ε, στο πλοίο και τη μείωση του κόστους για τους αλλοίς. Ε, προβλέπονται επίσης κάποιοι άλλοι κανόνες για μείωση των απορρίψεων. Ε, όπως για παράδειγμα ε, ένα καθεστώς παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται στη Βόρειο Θάλασσα. Επίσης, ε, πρέπει να δούμε ε, και ότι ε, θα εγκριθούν εδώ οι γενικοί, γενικοί κανόνες και στη συνέχεια οι επιμέρους κανόνες θα εφαρμοστούν μέσω επιτροπολογίας αποφεύγοντας τη μικροδιαχείριση σε, επίπεδο, σε γενικό επίπεδο πολιτικής. Όμως ορισμένες αστροπολογίες ζητούν κανονισμό του Συμβουλίου και για, τους, και για τα γενικά τεχνικά μέτρα αλλά και για τα επιμέρους τεχνικά μέτρα. Ιδιαίτερα όμως στα πλαίσια της μεταρρύθμισης κοινή ελευτικής πολιτικής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να εξακολουθήσει την μικροδιαχείριση ε, σε ε, γενικό επίπεδο Συμβουλίου. Ε, Πάντω η Επιτροπή είναι έτοιμη να, να μελετήσει πέραν τη Πετροπολογία οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα που θα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανέβει στο Συμβούλιο οποιοδήποτε ζήτημα θεωρούμε ότι είναι άκρος πολιτικό. Κυρίω είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τι τροπολογίε 2 και 3 που αναφέρονται ε, στις, ε, ε, στα, στα εργαλεία και ιδιαίτερα σε ορισμένε διατάξει αγορών, ιδιαίτερα όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθο των ειδών για, τον για την εναρμόνιση των μέτρων. Όσον αφορά τι απορρίψει, ε, η, Επιτροπή θέλει να ακολουθούν συγκεκριμένε διατάξει για, για ιδιαίτερε αλλίε με σκοπό τη μείωση των πρακτικών αυτών. Τα μέτρα αυτά θεωρούνται ότι είναι αποτελεσματικά εργαλεία και για να μειωθούν οι απορρίψει, αυτό το οποίο είναι ε, σημαντικό, ε, είναι να ε, επικεντρώσουμε ε, την προσοχή μας ε, στα αλλιεύματα και όχι στις εκφορτώσεις. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχθούμε ορισμένες από τι τροπολογίε σας που βαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όμως η τροπολογία 20 που θέλει να αντικατασταθεί, να χρησιμοποιηθεί το βάρος είναι αποδεκτή. Επίσης μπορούμε να θεωρήσουμε δεκτό και το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας όσον αφορά ορισμένες παρεκκλήσεις. Οι παράμετροι όμως αυτών των παρεκκλήσεων θα πρέπει να μελεχθούν στι λεπτομέρειε του και θα καθοριστούν στον εφαρμοστικό κανονισμό. Η Επιτροπή, ε, κυρίως για λόγους ε, ελέγχων, ε, θέλει να ακολουθήσει τον κανόνα του ενός δικτύου που θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερες περιπτώσεις. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε όμως για ιδιαίτερες περιπτώσεις αλίας εξαιρέσεις. Όμως με την προϋπόθεση ότι οι εξαιρέσεις αυτές είναι διόντως αιτιολογημένες και λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της τροπολογίας 11. Αυτές οι εξαιρεσει θα αποτελέσουν μέρος των περιφερειακών κανονισμών. Οι υπόλοιπε πτυχέ τη πρόταση επιτροπή είναι είναι άκρο τεχνικέ ε, και έχουν να κάνουν ε, με τη χρήση ε, των μέσων στον Ατλαντικό. Γνωρίζω ότι ο εισηγητή αλλά και η Επιτροπή Αλλία, ασχολήθηκαν με τα τεχνικά, τεχνικά τμήματα τη πρόταση και υπέβαλαν ορισμένε τροπολογίε με στόχο να είναι πιο αποτελεσματική η τροπολογία. Όσον αφορά όμω τι 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 και 22 τροπολογίε έχουμε επιφυλάξει. Γιατί εμείς προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε τις τεχνικές διατάξεις έτσι, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τον έλεγχο ε, στο ίδιο το πλοίο και να μειώσουμε το κόστος ε, των, ε, επί των αλλιέων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις 18 και 19 τροπολογίες γιατί υπήρξε ήδη πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθώντας τις επιστημονικές συμβουλές. Και, έχουμε τις, και, και, και απαιτούνται νέες, τεχνικέ πληροφορίε τεχνικές πληροφορίες για να τροποποιήσουμε τις διατάξεις αυτές. Δεν συμφωνούμε με την 27, με την τροπολογία 27. Βεβαίω θέλουμε να δώσουμε αρκετό χρόνο στου Ελλεί για να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε τεχνητό επίπεδο. Ε, για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρότασή του. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει ο κ. Καζάκα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Θέλω και εγώ να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την πρωτοβουλία νομοθετικού χαρακτήρα. Και επίση να συγχαρώ τον εισηγητή μα που εκπροσωπείται εδώ από την συνάδελφο Κάρμεν Φράγα. Θεωρώ ότι αληθεύει βέβαια ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κατεπήγον ε, κατεπήγοντα χαρακτήρα για την απλούστευση του νομοθετικού κώδικα σε σχέση με αυτά τα θέματα. Όμως πιστεύω ότι πρέπει ακόμα να πάμε αρκετά πιο πέρα σε δύο πράγματα κυρίως θεμελιώδου σημασίας. Το πρώτο είναι στα, στις απορρίψεις, στις απορρίψεις αλλιευμάτων. Στη μεταρρύθμιση που θα κάνουμε θα πρέπει να απαγορεύσουμε ως θέμα αρχής οποιαδήποτε απόρριψη. Θα πρέπει να απαγορευθούν κάθετα οι απορρίψεις και δεύτερον, θεωρώ ότι σε σχέση με την αρχή του σεβασμού των κανόνων που θα είναι περισσότερο αυστηροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλα τα σκάφη σε σχέση με τις περιοχές και περιφέρειες και τις αρμοδιότητες των περιφερειακών αρχών. Είναι δύο στοιχεία που πρέπει εδώ να ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη στην αναθεώρηση αυτή. Ευχαριστώ. κύριε Στο κυρία Ντόιλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τα μέτρα αυτά για επιλεκτικές πρακτικές αλίας ε, που θα βλάψουν στο δυνατόν λιγότερο τα περίπλοκα οικοσυστήματα και συγχρόνως θα επιτρέψουν τη συνέχιση μιας βιώσιμης ε, και λογικής αλίας ε, μείωση κατά το δυνατόν των απορρίψεων και αύξηση των εξόδων. Πράγματι πρέπει των εσόδων. Θα πρέπει σίγουρα το θέμα των απορρίψεων να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να δούμε επίσης πώς θα έχουμε την κατάλληλη επαρκή νομοθεσία, λαμβάνοντα υπόψη τις ιδιομορφίες και αναγνωρίζοντας ε, τη γνώση και την ε, εμπειρία των ε, επιτόπιων φορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητα. Είναι η τελευταία μας συζήτηση για την αλία σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε τόσο εσάς όσο και το προσωπικό σας ε, για την αφοσίωσή σας, ε, για τη βαθιά σας γνώση και για την προσοχή που δώσατε στην Επιτροπή μας ήσασταν πάντοτε διαθέσιμος ε, και πραγματικά ιδίω κάνοντας τη σύγκριση με άλλους επίτροπους και το πόσο διαθέσιμοι ήταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ο Επίτροπος. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ντόλ για τα πολύ ευγενικά της λόγια. Και να πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά τον κανονισμό αυτό, όπως ανέφερα και στην ε, πρώτη μου παρέμβαση, πράγματι η Επιτροπολογία θέλει ακριβώς αυτό να κάνει, να απλουστεύσει την ε, νομοθεσία πάνω σε πολύπλοκα ζητήματα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία που θα μας δώσει τη δυνατότητα παρόλα αυτά να θέτουμε ένα θέμα ε, στο Συμβούλιο, σε επίπεδο Συμβουλίου όταν είναι σημαντική η πολιτική διάσταση του θέματος. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να λαμβάνουμε μέτρα για τη μείωση των απορρίψεων, όπως είπατε, ιδίως ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, τις παραμέτρους της Βόρειας Θάλασσας και του σχεδίου του γάδου. Θα έχουμε και άλλες προτάσεις, παραδείγματο χάρη για το high grading και την κατάργησή του. Θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, για το 2010 και ελπίζουμε ότι μια ολιστική προσέγγιση και στο πλαίσιο και τη συζήτηση για τη μελλοντική ελευτική πολιτική να έχουμε ως τελικό αποτέλεσμα την οριστική εξάλληψη των απορρίψεων. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους ε, βουλευτές και δι' τα μέλη της Επιτροπής Αλίας για τη συνεχή υποστήριξη που έδειξαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που αφορούν την αλήθεια που τα οποία κάποτε ήταν ευαίσθητη. Κυρία Φράγκα, στέβες για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, κυρίως για κάτι το οποίο είπε, ότι είναι διατεθειμένος να ξαναδεί τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την Επιτροπολογία. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το Κοινοβούλιο μας σαφώς σε αυτή τη συζήτηση απέδειξε Στη συζήτηση δηλαδή στην Επιτροπή Ελία έδειξε ότι δεν συμφωνούμε με αυτή την πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αντικατοπτρίζεται και στο σχέδιο τη Πράσινη Βίβλου για τη μεταρρύθμιση κοινή ελευθερική πολιτική. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με αυτή την επιθυμία ε, ε, να να καταφεύγουμε εύκολα στην επιτροπολογία. Και το, τη δικαιολογία τη τάση τη αυτή η επιτροπή λέγοντα ότι τώρα απέναντι στη διαδικασία τη συναπόφαση, όπου το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά, μόλι αρχίσει να ισχύει και η συνθήκη τη Λισαβόνα, θα, ε, θα έχει αρμοδιότητε σε θέματα αλλία και φοβάται μήπω καθυστερήσουν οι διαδικασίε. Μα κοιτάξτε, δεν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι πολύ συχνά ε, καθυστερούν νομοθετικέ ε, ε διαδικασίε. Όχι ότι φταίει η διαδικασία τη συναπόφαση το Κοινοβούλιο, αλλά επειδή και η ίδια η Επιτροπή μερικέ φορέ καθυστερεί να υποβάλει την πρότασή τη. Γι' αυτό νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε και είναι ενδιαφέρον. Κατανοώ αυτό το οποίο είπε ο Επιτροπό, ότι σε ένα άκρο τεχνικό κανονισμό υπάρχουν ορισμένε τεχνικέ πτυχέ που πρέπει να αποφασίζονται μέσω επιτροπολογία και δεν μπορούν να περάσουν τα πάντα από το Συμβούλιο. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Επίτροπε, το θέμα είναι τι θεωρούμε τεχνικό, γιατί φαίνεται ότι εδώ υπάρχει διαφορά απόψε ανάμεσα σας και στο Κοινοβούλιο. Εμεί είμαστε πιο αυστηροί όσον αφορά το τι είναι τεχνικό και τι όχι. Δεν θέλω να επεκταθώ σε ένα θέμα, στο οποίο δεν ήμουν και συγγήτρια. Πάντω, σα πω το εξή, όσον αφορά τον κανόνα του ενιαίου δικτύου. Κοιτάξτε, ε, σε όλε τι συζητήσει που είχαμε στην Επιτροπή Αλία, αυτό το οποίο ξεκαθαρίστηκε είναι ότι η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή την αρχή κυρίω για λόγου ελέγχου. Όλοι βεβαίω συμφωνούμε ότι το θέμα αυτό, ε, ε ότι, ο έλεγχο είναι πολύ πιο απλό με ε, τον κανόνα αυτό. Αλλά ο κανόνα του ενιαίου δικτύου δημιουργεί προβλήματα σε ορισμένου αλληλευτικού τόλους, όπω το γνωρίζετε και εσεί πολύ καλά. Άρα λοιπόν, ε, μην κρυβόμαστε πίσω από τα θέματα του ελέγχου για να είμαστε πιο αυστηροί, όταν μερικέ φορέ δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα, ε, θα γίνει πληροφορία αύριο στις 12. Και τώρα θα περάσουμε στις έξι τελευταίες ε, εκθέσεις ε, της βραδιάς. Ε, συνάδελφοι, 10 λεφτά κατά μέσο όρο ανά έκθεση για να τελειώσουμε ε, στις 12. Γίνεται καταρχήν. Λοιπόν, σύντομη